Καλημέρα σας, καλό απόγευμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διακόψετε τις προσωπικές σας συζητήσεις. Κυρία Μπένα Ραμπατού, θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι πηγαίνετε στη θέση σας και καθόσαστε. Thank you very much. Ερχόμαστε στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. κύριος Σκουρία δυστυχώς δεν θα μπορεί να είναι παρόν αύριο το πρωί. Πρέπει να είναι παρόν στην ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και γι' αυτό μου ζήτησε το δικό του σημείο να προταχθεί και να εξεταστεί νωρίτερα. Η κυρία Κώστα έχει συμφωνήσει και αυτή. Θα αναστρέψουμε λοιπόν το 8 και το 9 αύριο. Σημείο 2 δεν υπάρχουν ε, τσέχικα, σλοβάκικα, λιθουανικά, λα... Ε, λετονικά, μαλτέζικα και είμαστε πάντα σε κατάσταση web streaming. Διαδιδόμαστε το διαδίκτυο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε ενώπιον μας την κυρία Νέιλι Κρούς, η οποία είναι αρμόδιος επίτροπος για το θεματικό, για το ψηφιακό θεματολόγιο στις τέσσερις. 4 και 4 πρέπει να φύγει η κυρία Επίτροπος, γιατί στις 4.30 συναντώνται οι Υπουργοί Αθλητισμού και Πολιτισμού, που ήταν αγίτη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω της διάσκεψης κορφής έχει μεταφερθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω αμέσως το λόγο. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πήρατε ξανά την πρωτοβουλία να με καλέσετε εδώ στην Επιτροπή σας ώστε να σας ε, ενημερώσω για το έργο μας. Είναι σαφές, δεν είναι νέο αυτό που θα σας πω. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύσκολες εποχές, αναμφίβολα, απασχόληση, ύφεση, απώλεια ανταγωνιστικότητας. Οι δημιουργικές βιομηχανίες και το πολιτισμικό περιεχόμενο έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κομμάτι της λύσης κατά κάποιο τρόπο, διότι ο πολιτισμός βοηθάει την κοινωνία μας, υποστηρίζει την ένταξη όλων των ομάδων, την εκπαίδευση και τη δημοκρατική ελευθερία. Υποστηρίζει όμως επίσης, κυρία Πρόεδρε, και την οικονομία μας σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν λίγο παραπάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα, αν μου επιτρέπετε, ήθελα να μιλήσω για τρεις ε, τομείς του χαρτοφυλακίου μου που έχουν ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας και θα ζητήσω και τις απόψεις για τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, πώς ε, εναγκαλίζοντας το διαδίκτυο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ε, ε, τομέα για την ευημερία. Δεύτερον, πώς υποστηρίζουμε την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, πώς χρειαζόμαστε υποδομέ, ψηφιακέ και πλαίσια ώστε να γίνουν όλα αυτά. Πολλέ πτυχέ λοιπόν τη ζωής μας, όλο και περισσότερο, περνούν στο διαδίκτυο ψυχαγωγία, πολιτισμός, δημιουργικότητα. Α θυμηθούμε τις ευκαιρίε και τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάσταση για τον τομέα του πολιτισμού. Το έχουμε συζητήσει για παράδειγμα ε, το να έδειξε τεράστιες δυνατότητες ε, ευρείας πρόσβεσης σε ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες προσπάθειες ώστε να αυξήσουμε το προσπελάσιμο περιεχόμενο. Ακόμα συμβαίνει κάποιοι άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό. Κάτι άλλο, η κινηματογραφική κληρονομιά είναι ένας τομέας όπου απομένουν να γίνουν πολλά η τρίτη μας ε, έκθεση υλοποίηση που θα κυκλοφορήσει σύντομα θα δείξει ότι το 85% της κινηματογραφικής κληρονομιάς της Ευρώπης είναι εκτός εμπορίου συνεπώς μη προσπελάσιμο ενώ το 98,5% δεν έχει ψηφιοποιηθεί. Παραμένει κλειδωμένο σε αυτές τις μεταλλικές θήκες ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται online και προσπελάσιμο σε όλους μας. Όσον αφορά τα βιβλία, συμβαίνει το ίδιο τον Ιούνιο φέτος. Ε, συναντήσαμε σημαντικούς παράγοντες ε, της αλυσίδας αξίας βιβλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουμε ευκαιρίες και εμπόδια για τον τομέα. Οι παρόντες ε, υποστήριξαν την αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχουν φραγμοί στην αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων ε, διασυνοριακά και σε όλα τα είδη συσκευών. Αυτό θα ήταν μια επανάσταση για τα ηλεκτρονικά βιβλία και για την ενιαία μας αγορά. Κοιτώντα τον οπτικοακουστικό τομέα, ευχαριστούμε τον κύριο Μπόρι για την έκθεσή σας για την οδηγία AVMS. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, ενώ προστατεύει σημαντικού στόχου πολιτική όπω την προστασία των παιδιών. Αλλά τα οπτικοακουστικά μέσα και αυτά περνούν στο διαδίκτυο και μετατρέπονται οι συσκευές που συνδέουν το ίντερνετ με τις ε, εκπομπές ε, εξαπλώνονται ταχύτατα σε τηλεοράσεις, σε έξυπνα τηλέφωνα και εμείς ε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις τεχνολογικές και επιστημονικές και ίσως και νομικές συνέπειες. Πράγματι σχεδιάζουμε μια πράσινη βίβλο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση για τις αρχές του επόμενου έτους. ορίζω ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας γενικότερα, καθώς και την εκθέση Κάμερβερτ. Γενικώ το διαδικτύο αλλάζει όλο τον τομέα των μέσων μαζική ενημέρωση και εμεί δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτή την αλλαγή. Αλλά αν δεν κάνουμε τα πράγματα σωστά, θα μείνουμε πίσω σε σχέση με τους παγκόσμιους εταίρους μας προς απώλεια των πολιτών μας, της δημοκρατίας μας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, του ευρωπαϊκού τομέα μέσων ε, μαζική ενημέρωση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τις προκλήσεις αυτές. Αυτό είναι το μήνυμα τη έκθεση που μου το φόρουμ ε, μελλοντικών μέσων του κυρίου Κριστιαν Βαντήλο. Εκεί γίνονται διάφορε συστάσει για το πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Παρεμπιπτόντω, ε, ήταν η μόνη ομάδα όπου σε όλη μου την ενεργό επαγγελματική ζωή ρωτούσαν κατά πόσο είναι αποδεκτό να παρουσιαστεί μια έκθεση νωρίτερα από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Για παράδειγμα, μιλάω για τις συστάσεις του φόρουμ με την ευθυγράμμιση των ΦΠΑ online και offline ή νέων συστημάτων μικροπληρωμών, ώστε να είναι ευκολότερο να πληρώσει κανείς για περιεχόμενο online, ακόμη και αν πρόκειται για ένα μόνο ευρώ και γνωρίζω ότι ο κύριος Φαντήλο σκοπεύει να μιλήσει με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβάνεις και της Δικής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τις συστάσεις του. Το ερώτημα μου λοιπόν εδώ προς όλους σας είναι πώς θα οικοδομήσουμε το σωστό πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει τον τομέα στην ψηφιακή εποχή. Πώς για παράδειγμα μπορούμε να αιτιολογήσουμε ότι θα πληρώνετε χαμηλότερους φόρους για να αγοράσετε μια ε, ψηφιακή, μια εκτυπωμένη εφημερίδα από ότι να κατεβάσετε μια εφημερίδα από το διαδίκτυο. Μιλάμε τώρα για καθημερινή βάση. Τι προτιμάτε, την εφημερίδα την ίδια ή να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλέον αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι ο υπολογιστής. Πώς μπορούμε να αιτιολογήσουμε λοιπόν ότι θα πληρώνει κανεί χαμηλότερο φόρο για την έντυπη έκδοση από ότι για την ψηφιακή λήψη μια εφημερίδα. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό σε, σε πολλού ανθρώπου. Είναι το ίδιο περιεχόμενο, διαφορετικά ΦΠΑ και αφορά το περιεχόμενο, όχι τη φόρμα. Δεν πληρώνει περισσότερο ΦΠΑ για ένα δώρο εάν το τυλίξεις με χρυσό ή με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Από την άλλη γνωρίζω ότι πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής ε, γνωρίζουν και μελετούν τα θέματα των διανοητικών δικαιωμάτων και των παραβιάσεων. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να εξυπηρετεί τους δημιουργούς αλλά το θέμα είναι ότι οι πιο σκληρές δράσεις δεν είναι βιώσιμες. Το είδαμε και στην περίπτωση της Άκτα. Πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από τα όσα έγιναν σε σχέση με την άκτα στην οποία εσείς δραστηριοποιηθήκατε ιδιαίτερο και πιστεύω είχατε δίκιο. Θα πρέπει λοιπόν να αποκομίσουμε τα διδάγματα από αυτό το τομέα. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση περιεχομένου online νόμιμα, να κάνουμε το σύστημα προστασίας διανοητικών δικαιωμάτων κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή και πώς μπορούν οι καλλιτέχνες μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους προέρχονται online. Επίσης πώς θα μπορέσουμε να υπερασπίσουμε την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι ζητήματα που θέτω με πολύ ε, ισχυρούς όρους στην πρόσφατη επισκέψη μου στον Πακού του Αζερμπαϊτζάν. Το ίδιο έπραξα και στη συναντησή μου με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν. Η ελευθερία λόγου είναι ένα πολύτιμο ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω στη δική σα επιτροπή. Είναι μία από τις κυριότερες αρχές μιας δημοκρατίας. Επίσης όμως και η ελευθερία μετά τον λόγο είναι σημαντική. Και αυτό σαφές μετά την επισκέψη μου στο Αζερμπαϊτζάν ότι ε, πίνουμε ε, διαφορετικό τσάι, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Όταν κάποιο καταδιώκεται επειδή τολμάει να μιλήσει, τότε δεν υπάρχει ελευθερία ομιλία. Και ευχαριστώ τα μέλη τη Επιτροπή αυτή που συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη και βοήθησαν στη διεξαγωγή τη. Το ζήτημα τη ελευθερία των μέσων δεν είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο χαρτοφυλακιό με το ψηφιακό θεματολόγιο. Σχετίζονται απολύτω. Είναι σαφέ ότι το διαδίκτυο είναι μια νέα μορφή, ένα νέο σύνορο ελευθερίας επιτρέπει τον πλουραλισμό και ας θυμηθούμε πως ένα κορίτσι εξοπλισμένο μόνο με μια διαδικτυακή σύνδεση κατάφερε να αντισταθεί στο Ταλιμπάν και να διαδώσει ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά η ελευθερία και ο πλουραλισμό των μέσων αποτελούν ζητήματα και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει πολλέ εξέξω περιπτώσει στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία αλλά ουσιαστικά αποτελεί ένα ζήτημα που τίθεται σε πολλά κράτη-μέλη. Ας κοιτάξουμε την όλη συζήτηση ε, Λέβεσον στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την πρόσφατη σύλληψη ενός δημοσιογράφου στην Ελλάδα ή στην εκπομπή δημοσίων υπηρεσιών στην Πορτογαλία. Πώς θα ανταποκριθούμε, πώς θα αποκριθούμε. Έχουμε κάποια εργαλεία. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας χρησιμοποίησαμε εξουσίες δυναμή της ε, οδηγίας AVS και μπορούμε να εξασκήσουμε πολιτική πίεση όπως έκανα πρόσφατα στη Βουλγαρία. Δεν δίστασα να το πράξω τότε και δεν θα ξαναδιστάσω στο μέλλον εφόσον χρειαστεί. Διότι το θέμα εδώ είναι η αξιοπιστία. Μας κατηγόρησαν στον Πακού, στο Ζαρμπαϊτζάν ότι δεν είμαστε δίκαιοι προς αυτούς ε, αν δεν κάνουμε το ίδιο και στην Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία μετά τον λόγο, τότε πρέπει να το πράττουμε παντού. Διότι... Τώρα, η πολιτική πίεση χωρί επιβολή του νόμου είναι επαρκή. Εδώ οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένε και εμεί γνωρίζουμε σε μια παλιότερη συζήτηση, κατά τη συζήτηση για την Ουγγαρία, διαπιστώσαμε τους περιορισμούς σε σχέση με τα διακυβεύματα και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο, ο τρόπος υποστήριξης της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Ένα από τα κυριότερα αφορά το θεμελιωδή λίθο μιας δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο ο καθηγητής Φάιρεφικα Φρέιμπεργκα θα παρουσιάσει τις διαπιστώσεις της δικής της ομάδας υψηλοεπέδου για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για μια ευρύτερη συζήτηση. Επαναλαμβάνοντας λοιπόν την ερώτησή μου προς εσάς και την ερώτηση που έκαναν νωρίτερα φέτος, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα σε αυτό το τομέα. Αν ναι, από ποιον και χρησιμοποιώντας ποια εργαλεία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συμβολή και τη συνεισφορά της Επιτροπής μέχρι σήμερα. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση με όλους σας, με τους ενδιαφερόμενους, με τα κρατημέλη, ώστε να ε, αποφασίσουμε κάποιον τρόπο για το μέλλον πριν από το τέλος εντολής της Επιτροπής Μπαρόσο. Το τρίτο σημείο σήμερα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο με ένα πιο γενικό τρόπο. Ένα τρόπο υποστηρίξη των δημιουργικών τομέων είναι να εξετάσουμε τον κάθε δευτερεύοντα τομέα, κινηματογράφο, βιβλία, τηλεόραση, ξεχωριστά. Αλλά αυτό, κατά την άποψή μου, δεν αρκεί κατά πολλού τρόπου. Ο καλύτερο τρόπο να δημιουργήσουμε το δημιουργικό τομέα είναι να παρέχουμε ψηφιακή υποδομή, δίκτυα και πλαίσια που υποστηρίζουν την ψηφιακή κοινωνία. Και επειδή η παροχή αυτής της ε, υποδομής ε, θα βοηθήσει στην καινοτομία, ε, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί τόσο αυτόν τον τομέα όσο και σε άλλους. Φανταστείτε για παράδειγμα κυρίε και κύριοι, εάν οι αγαπημένες σας ταινίες, τα αγαπημένα σας βιβλία, η αγαπημένη σας μουσική είχαν αποθηκευτεί κάπου σε ένα μου κάπου όπου θα είχατε πρόσβαση εκεί νόμιμα, άμεσα, εφόσον το ζητήσετε μέσω γρήγορου δικτύου όπου και να βρίσκεστε και όποια συσκευή και να χρησιμοποιείτε φανταστείτε τι πλεονέκτημα θα ήταν κάτι τέτοιο για τη δημιουργική μας βιομηχανία και για τους πολίτες μας. Διότι τότε η ψηφιακή ενιαία αγορά θα αποτελούσε κάτι πραγματικά σημαντικό για τους πολίτες. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό ζήτημα. Το φόρουμ για το μέλλον των μέσων κατήστησε σαφές ότι η γρήγορε ευρυζωνικέ συνδέσει είναι ουσιώδη σημασία για να υποστηρίξουν τον τομέα των μέσων. Συμφωνώ και εγώ και θα το πρόσθετα και για οποιοδήποτε άλλο τομέα. Διότι μακροπρόθεσμα και για αυτό το ε, ευρυζωνικό δίκτυο χρειαζόμαστε και πλαίσια να έρουμε του φραγμούς για το υπολογιστικό νέφος να δώσουμε μια νέα κατοικία για την δική μας ενία αγορά και ένα πλαίσιο για την προστασία των παιδιών ώστε τα παιδιά να μπορούν να διασκεδάζουν με ασφάλεια online. Και πράγματι μετά από αυτή τη συνάντηση εδώ θα παραστώ στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης Νέων και Πολιτισμού που θα ζητήσουμε ακριβώ αυτό το ζήτημα. Καθώς και ένα πλαίσιο όπου θα είναι ευκολότερη η ασφαλής πρόσβαση σε περιεχόμενο online αξιοποιώντα όλα τα ωφέλη της νέας ψηφιακής μας αγοράς. Η οδηγία μας που προτείνει μεταρρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης αποτελεί σημαντικό ζήτημα, αλλά έχουμε και άλλα ζητήματα επίγοντα να αντιμετωπίσουμε, όπως το να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε οπτικοστικά μέσα online, συμπεριλαμβανομένης και τη διασυνοριακή διάστασης και να φτιάξουμε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο copyright, λιγότερο κατακαιρματισμένο. Σε λιγότερα από δύο χρόνια θα ανα θα δημοσιεύσουμε την ε, ανασκόπηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρωπαϊκή και πρέπει να σας δηλώσω ότι έχει σημειώσει τεράστιες πρόοδους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχουν αυξηθεί η χρήση του δικτύου από μειονεκτούς ομάδας και οι αγορές online. Το 95% των οικειών στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν σταθερή ευρυζωνική σύνδεση διαθέσιμη και όλο και περισσότεροι έχουν πρόσβαση σε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, ενώ το 50% των κατοικιών έχουν πρόσβαση σε υψηλή ταχύτητα κάλυψη. Όλο και περισσότερο οι Ευρώπαιοι διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα των ταχύτερων συνδέσεων. Οι συνδρομέ αυτέ αυξάνονται. Η ανασκόπησή μα του ψηφιακού θεματολογίου θα επανεστιαστεί σε ορισμένου τομείς κλειδιά που είναι απαραίτητοι για την τόνωση της ψηφιακής μας οικονομίας. η ε, υψηλή ευρυ, ε, ζωνική σύνδεση, ε, υπολογιστικό νέφος, περιεχόμενο online, online υπηρεσίες και έρευνα και ανάπτυξη. Για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη προτείναμε να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά πρώτα εξασφαλίζοντας ιδιωτική χρηματοδότηση ώστε 45 εκατομμύρια οικίες να συνδεθούν σε ταχύ ευρυζωνικό δίκτυο μόνο φέτος το 2012 στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 36 εκατομμύρια οικίες θα συνδεθούν με ταχύ ευρυζωνικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επιταχύνουμε και να διασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά όταν υπάρχουν οι υποδομές τότε και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει και τις πολιτιστικές υπηρεσίες όπως το Ευρωπαϊκό. Ελπίζω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι το Κοινοβούλιο σας και η δική σας Επιτροπή θα υποστηρίξει την πρόταση για το μέσο αυτό και θα αναγνωρίσουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ψηφιακή ανάγκη και σε αυτήν την ψηφιακή πρόκληση θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Το τρίτο ερώτημα που θέτω λοιπόν, το τελικό σήμερα, ε, για να ληφθούν οι αποφάσεις είναι το πώς θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να τους δείξουμε ότι εμείς έχουμε μπροστά μας μια οικονομικά ε, σημαντικότατη επένδυση σε μια δημιουργική βιομηχανία ε, εφόσον πραγματικά λειτουργήσουμε σαν Ήπειρος η οποία θα είναι ψηφιακά συνδεδεμένη. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ήταν πραγματικά πολύ σύντομα. Ελπίζω ότι έχουν περάσει ώρα στη διερμηνία. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε εσείς Έχετε φυσικά και την υποστήριξη της κυρίας Βασιλείου και άλλων επιτρόπων. Όλα για αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Χέσου έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχουμε πολύ συναρπαστικά θέματα στην ημερήσια διαταξή μας, τα οποία εν μέρει αναφέρατε και εσείς. Έχω δύο ερωτήματα για εσάς. Το πρώτο ερώτημα, σε σχέση με την ε, πρωτοβουλία για τη συνδεδεμένη τηλεόραση. Υπάρχουν ορισμένα κεντρικά σημεία τα οποία εμεί έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα παίξει τον κύριο ρόλο. Είναι ο πάροχο υπηρεσία, ο οποίο θα αφήσει το περιεχόμενο που θέλει, είναι ο κατασκευαστής ο οποίο θα αποφασίσει και έχουμε τελικά το θέμα της προστασίας των νέων από την, από την διαφήμιση και το βλαβερό περιεχόμενο για τους νέους και τους εφήβους. Πώς θα συνεργαστείτε λοιπόν με του υπόλοιπου επιτρόπους για το θέμα αυτό πώς θα προχωρήσουν αυτά τα, θέματα και θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα μέχρι τις ευρωεκλογέ του 2014. Και αν εμείς έχουμε αβεβαιότητα για τα θέματα αυτά, για τον δημιουργικό τομέα του οπτικοακουστικού, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και δεν μπορούν να σχεδιάσουν σωστά τις ενέργειές τους. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά την Ουγγαρία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ουγγαρία σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία των ε, μέσων ενημέρωσης, υπάρχει περιορισμός και καταστολή τους από τις ε, πολιτικές αρχές. Κυρία Σάντσεθ Σμιτ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την δέσμευσή της για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη στα ψηφιακά θέματα Νομίζω ότι ο κάθε Ευρωπαίος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες οι οποίες, οι οποίες ανοίγουν τόσες δυνατότητες σε όλους τους πολίτες μας. Έτσι μπορούμε λοιπόν να απελευθερώσουμε και την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά έργα τέχνης, αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊάνα, να υπάρχει πρόσβαση στο οπτικό-ακουστικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες να κατανοήσουν και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια είχαμε ψηφίσει την έκθεση της κυρίας Κώστα για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό χώρο. Χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία θα προσαρμόσουν καλύτερα τη χρήση του διαδικτύου στα παιδιά και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παροτρινθεί η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και μια καλύτερη υποστήριξη στην ψηφιακή οικονομία, κυρίως με την καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών στα οπτικοακουστικά θέματα. Συγχρόνως, όπως είπαμε, πρέπει να υπάρξει η καλύτερη προστασία πάντα μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των ε, οπτικοακουστικών δημιουργών. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα θέματα του σεβασμού των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Το δείξατε αυτό σε σχέση με τα δικαιώματα στον επιγραμμικό χώρο. Αυτά ποικίλουν από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δημιουργηθούν και ελλείψεις ισορροπίας όταν κάποιος τομέας μπορεί να αποκτήσει ένα μονοπόλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε τα ψηφιακά θέματα. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και την απαραίτητη προσαρμογή που χρειάζεται λόγω της πολυγλωσσικότητας της Ευρώπης. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η πολυμορφία, η γλωσσική και η πολιστική είναι μια δύναμη για την Ευρώπη, είναι πηγή ε, πλούτου για την Ευρώπη και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ρωτήσατε κύριε Επίτροπε τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Νομίζω ότι η Ευρώπη απαιτεί μια μεγαλύτερη προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε όλους. Πώς θα βρούμε λοιπόν τα πώς θα εντοπίσουμε τα εμπόδια και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε. Έχουμε τα νομοθετικά εργαλεία, αλλά επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε και εργαλεία για να προωθήσουμε τα προγράμματα και στην Επιτροπή μας εργαζόμαστε για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μέχρι το 2020 και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε πράγματι να παρακολουθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια για καλύτερη προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστώ. κυρία Κάμερφερτ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο, την κυρία Κρούς για τα λόγια της. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το θέμα της συνδεδεμένης τηλεόρασης, γιατί δυστυχώς δεν θα είναι εδώ η Επίτροπος όταν εγώ παρουσιάσω τις πρώτες μου σκέψεις για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα είναι χρήσιμο για μένα η Κομισιόν να προετοιμάσει μια πράσινη βίβλο για τα θέματα αυτά, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην καθυστερήσετε πάρα πολύ για το να προτείνετε μέτρα για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ρευστέ οι συνθήκε, υπάρχει πολύ ταχεία εξέλιξη και εμεί ω πολιτικοί πάντα κινδυνεύουμε να υπολοιπόμαθα πολύ τη τεχνολογική εξέλιξη. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι γίνεται εκ, του, εκ των πραγμάτων υπάρχει μια εξέλιξη που οδηγεί σε κανονιστικά και ρυθμιστικά μέτρα και είναι απαραίτητο εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να φέρουμε τις κατάλληλες ρυθμίσει για τα θέματα αυτά και να μην αφήσουμε τα de facto πρότυπα να επιβληθούν για να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια για το μέλλον. Και είπατε πολλά για την ε, ελευθερία του διαδικτύου και με ικανοποιεί αυτό. Θα ήθελα να σας επιθυμίσω και πάλι το ψήφισμα το οποίο ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την επικείμενη συνδιάσκεψη του Ντούμπαϊ για τα θέματα επικοινωνιών, όπου ε, εμείς θέλουμε να εφέρουμε τις δικές μας ανησυχίες ως Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι από τη Ρωσία αλλά και από τα αραβικά κράτη που θέλουν να υπάρξει σημαντικός περιορισμός της ελευθερίας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό, κύριε Κρούς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω μαζί με τους συναδέλφους σας και μαζί με τα κράτη-μέλη τα οποία είναι και αυτά οι, τα συμβαλόμενα μέρη στην διάσκεψη του Ντουμπάι να καταβάλλεται τις απαραίτητες προσπάθειες για να διατηρηθεί η ελευθερία του ίντερνετ. Νομίζω ότι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούμε να προωθήσουμε μια ρύθμιση και έχουμε κάνει σαφές στο δικό μας ψήφισμα ότι δεν θα αποδεχτούμε σε διεθνές επίπεδο περιορισμούς της ελευθερίας του ίντερνετ. Ελπίζω ότι και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη με τη δική σας παρότρινση θα πάρουν τις σωστές θέσεις, ώστε από την συνδιάσκεψη του Ντουμπάι θα προκύψουν λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές για την Ευρώπη και όλους μας. Είπατε ότι έχουμε μάθει το μάθημά μας από, το, από τα, τη διαδικασία του νομοθετήματος ΑΚΤΑ. Νομίζω ότι πράγματι αυτό ελπίζω ότι πρέπει να είναι πραγματικότητα. Υπάρχει μια σαφή στάση η οποία διατυπώθηκε και την εποχή του Άκτα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ίντερνετ δεν θα ελέγχεται με τρόπο ο οποίος θα είναι περιοριστικός. Δεν πρέπει οι τρόποι με τους οποίους θα ρυθμίσουμε το ίντερνετ να οδηγήσουν στη μείωση ε, των βασικών ελευθεριών μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και το δικαίωμα έκφρασης που είναι από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης δεν πρέπει να θυγεί η πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης. Το θέμα λοιπόν είναι σε ποιο βαθμό εμείς πρέπει να ελέγχουμε τις ροές πληροφορίες από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχει ένας ε, χώρος ελευθερίας που μας δίνει το ίντερνετ, θα πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό τον χώρο ελευθερίας και θα πρέπει να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία για την προστασία των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, ώστε και να έχει ο πνευματικός δημιουργός το δικαίωμα να απολαμβάνει την, της ιδιοκτησίας του, αλλά και ο καταναλωτής και ο χρήστης του ίντερνετ να μην υπόκειται σε υπερβολικούς περιορισμούς, ώστε και να χάνει και κάθε ενδιαφέρον να αναζητεί όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέλει να μάθει στο διαδίκτυο. Δεν πρέπει λοιπόν να απορρίπτουμε το βρέφος με τα ύδατα κολύμβησης του ιδίου αυτού βρέφους. Ό,τι ελέγχθη επίσης για την πρόσβαση στο ακουστικό περιεχόμενο ε, ε, online, επιγραμμικά. Εμεί έχουμε προσπαθήσει να προχωρήσουμε με την ε, οδηγία για τα ορφανά έργα, καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ήταν, πιστεύω, ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν ήταν αρκετά θαραλέο αυτό το βήμα σε σχέση με τα οπτικοακουστικά έργα. Εδώ παραμένουν πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά εμπόδια για τα πολλά αυτά έργα, τα οποία βρίσκονται και μαζεύουν σκόνη σε κάποιο αρχείο στα κράτη-μέλη μας, γιατί υπάρχει δυσκολία να μπορέσουμε να τα ψηφιοποιήσουμε. Αυτό με τις τωρινές ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τουλάχιστον αυτή η οδηγία θα πρέπει να βοηθήσει τα ορφανά έργα ή τα εν μέρη ορφανά έργα να μπορέσουν να έρθουν στην ε, δημοσιότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο λοιπόν και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω να εξ αρχής για την θέλησή σας να λάβετε υπόψη και τη ρήτρα αναθεώρησης για αυτή την οδηγία. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης, ώστε όταν γίνει αυτή η αναθεώρηση να προχωρήσουμε με πιο θαραλέα βήματα, ώστε αυτή η καλλιτεχνική θησαυρή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορα αρχεία να μπορέσουν να έρθουν στο προσκήνιο και να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν προσβάσιμε στο διαδίκτυο αυτή η καλλιτεχνική θησαυρία. Αυτό θα έχει προωθήσει ιδιαίτερα την πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη. Κυρία Πατού. Ε, Ευχαριστώ Επίτροπε. Ευχαριστώ για το πανόραμα το οποίο μας παρουσιάσατε. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και σε πολλούς τομείς. Μία από τις βασικές ερωτήσεις αφορά την χρηματοδότηση των εφημερίδων. Μιλήσατε για τις εφημερίδες σε χαρτί, για τις εφημερίδες στο διαδίκτυο. Πώς προβλέπετε τη χρηματοδότησή τους. Δύο υπάρχουν δυνατότητες. Ή η χρηματοδότηση μέσω διαφημίσεων αλλά με μεγάλη εξάρτηση από τις εταιρείες και από τις διαφομιστικές εταιρείες είτε από το σύστημα των συνδρομών. Πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα το δικό σας όραμα σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των νέων μέσων, τα οποία θα ε, λειτουργήσουν πλέον κατά πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται στο μέλλον. Τώρα, ο δημοκρατικός χαρακτήρας αυτών των νέων μέσων. Επιμείνω εδώ στη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Ζούμε σε ένα κόσμο που όταν ξεκινήσαμε δεν ήταν ο πιο σημαντικός κόσμος ο ψηφιακός. Πρέπει να εκπαιδευτούμε λοιπόν. Μιλήσατε επίσης και για την ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί αλλιώς ο κινηματογράφος δεν θα είναι για όλους διαθέσιμος. Ε, τι είδους χρηματοδότηση θα υπάρξει. Αυτή η ψηφιοποίηση θα κοστίσει πάρα πολύ αν θέλουμε πραγματικά να καταστεί διαθέσιμη κληρονομιά σε όλους τους πολίτες. Τέλος, για τη συνδεδεμένη τηλεόραση, πάρα πολύ σημαντικό και δημοφιλές οικογενειακό μέσο. Η τηλεόραση αυτή θα ανατρέψει τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο λειτουργίας τους. Έμαθα με χαρά ότι μια πράσινη βίβλος θα δημοσιευθεί τάχιστα επί του θέματος. Γνώμη δική σας ποια είναι για τα χαρακτηριστικά αυτής της συνδεδεμένης τηλεόρασης, η οποία θα είναι τελικά η νέα τηλεόραση για τα επόμενα χρόνια. Και τέλος, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα πνευματικά δικαιώματα, μετά από την καταπλειοψηφία ψήφο του Κοινοβουλίου εις βάρος του ΑΚΤΑ, της Συμφωνίας ΑΚΤΑ, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τα πνευματικά δικαιώματα. Μιλήσατε για τον εξυγχρονισμό των δικαιωμάτων αυτών. Πώς θα γίνει, σε ποια βάση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακαλάρκινα. Ευχαριστώ κύριε Πετρόπα. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ήθελα να σας δω και στη Washington για την παγκόσμια σημασία για την προστασία των παιδιών, αλλά ο τυφώνα Σάντι σας εμπόδισε. Αλλά θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν γίνεται τι γίνεται σήμερα όσον αφορά την προστασία των παιδιών online. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το παρακολουθούμε και ότι θα καταφέρουμε να το επιτύχουμε αποτελεσματικά. Ήθελα να μα πείτε τι κάνετε σε αυτόν τον τομέα. Το ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο ασχολείστε, καλύπτει πολλέ γενικέ διευθύνσει και πολλέ επιτροπέ και εδώ νομικέ ε, αγορά. Και πραγματικά εκτιμάμε που βρίσκεστε εδώ ώστε να μα βοηθήσετε να υπερασπίσουμε και τι πολιτισμικέ μα αξίε. Έχουμε πολλά θέματα φυσικά αλλά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πλαίσιο για το copyright, με τα πραγματικά δικαιώματα. Θέλαμε να μας πείτε πώς εξελίσσεται. Ουσιαστικά τελειώνει ο χρόνος, ε. φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της εντολής και πολλοί τομείς ε, ε, που περιλαμβάνουν το copyright ως θέμα θα χρειαστεί να επιταχύνουν. Κοιτώντας αυτό, όπως και το AVMS, θέλουμε να δούμε τι είναι νομικά δυνατό, αλλά και τι είναι τεχνικά δυνατό. Δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε και την τεχνική πτυχή των πραγμάτων, για να παρακολουθούμε και την τεχνολογία. Ουσιαστικά είναι ένα αγώνα το να προσπαθούμε να καταλάβουμε την τεχνολογία πάνω στην οποία εργαζόμαστε και θα θέλαμε να μα συμβουλέψετε γι' αυτό τώρα όσον αφορά το EVMS, όσον αφορά την υλοποίηση του EVMS, τα όσα μαθαίνουμε από αυτή την υλοποίηση. Θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε μπροστά καθώς θα κάνουμε την ανασκόπηση διότι ξέρω ότι σε κάθε κράτος μέλος υλοποιήθηκε διαφορετικά και ήθελα να μου πείτε πώς θα συνδεθεί αυτό με την Connected TV. Χαίρομαι για την εξέλιξη του πολύ γρήγορου ευρυζωνικού δικτύου αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αφορά κυρίω τις πόλεις και όχι τι αγροτικέ περιοχέ. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα για μένα και στην περιοχή μου. Ευχαριστούμε και για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά ήθελα να μου πείτε τι θα κάνετε ακριβώ ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτά τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλή ταχύτητα. Ευχαριστώ. Κώστα. Κυρία Κώστα. Σίλβια. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επιθυμία σας να συλλέξετε προτάσεις, ιδέες και ευαισθησίες από την Επιτροπή μας πάνω στα θέματα που θέσατε και τα οποία είναι θέματα τα οποία κινούνται και αλλάζουν συνεχώς. Χαίρομαι που υπήρξε συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των ανηλίκων καταρχάς στον ψηφιακό κόσμο. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της πρόσφατης συμφωνίας που υπογράψατε με τη ΣΥΠΑ για τη συμμετοχή και τον ΗΠΑ στο Safer Internet, τη διεύρυνση της ε, σφαίρας ευθύνης γύρω από τα θέματα αυτά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και εδώ εγγράφεται και η οδηγία της κυρίας Ρένινγκ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία σας και μετά από την πρόσφατη ανακοίνωσή σας, η οποία όπως είπα συμπίπτει με τη δική μου έκθεση. Το θέμα των ανηλίκων βέβαια δεν θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε, πρέπει να κάνουμε και κάποια επιπλέον βήματα στα πλαίσια της οδηγίας για τις τηλεοπτικές υπηρεσίες που δεν καλύπτει όλες τις επιγραμμικές μορφές επικοινωνίας. Κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν και άλλα θέματα, όπως σαν παράδειγμα η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξέρουμε ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή, η μεγάλη αυτή αλλά και η ψηφιοποίηση γενικότερα της κινηματογραφικής κληρονομιάς. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε η ψηφιοποίηση είναι αρμοδιότητα κυρίως ε, δική σας. Είναι στο χαρτοφυλάκιό σας και καλύπτεται και από τα διαφθορτικά ταμεία. Οπότε πώς ακριβώς θα πρέπει να παραπέμψετε το θέμα αυτό και σε άλλες νομικές βάσεις για την ε, προοδό του. Όταν το Κοινοβούλιο σε ένα πρόσφατο ψήφισμά του του 2011 ε, ζήτησε να μάθει γιατί υπάρχει μια ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό για την ψηφιοποίηση για την πνευματική κληρονομιά, η απάντηση που είχατε δώσει είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά των κρατών μελών. αλλά ο κανονισμός πράγματι λέει στο άρθρο 4 ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Θα πρέπει όμως να δούμε ε, τι γίνεται με την έννοια ψηφιοποίηση. Εδώ δεν τίθεται καθόλου η έννοια αυτή. Ε, ποιος είναι υπεύθυνο για να στηρίξει την ψηφιοποίηση. Δεν θα ήθελα ο ένας να τα ρίχνει στον άλλο και να μην αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες του. Τελευταία παρατήρηση το θέμα της ε, υποχρεωτικής παρέμβασης στην περίπτωση που υπάρχει σαν πραγματικά διαφορετική, μεγάλη διαφορά στο κόστος πρόσβασης στο ευρύ φάσμα και στο ψηφιακό περιεχόμενο με ενιαίο τρόπο. Θα πρέπει να το δούμε και λίγο ανάποδα αυτό βέβαια. Υπάρχουν χώρες εδώ οι οποίες ακολουθούν διαφορετικές γραμμές. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη ανησυχία όμως κυρίως από πλευράς ε, των δημιουργών και των πνευματικών δημιουργών. Οι παροχή εκπομπών σαν παράδειγμα και υλικού ψηφιακού δεν σέβονται πάντα τους κανόνες. Ε, δέχονται κυρίως και σέβονται το λεγόμενο value chain, την αξία την εμπορική του προϊόντος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε χρεώσεις απαράδεκτες οι οποίες ε, δεν είναι θα έλεγα ε, νόμιμες και δεν υπάρχει επιστροφή και αποζημίωση των παραγωγών αυτών που ήταν υπεύθυνοι για την παραγωγή του συγκεκριμένου περιεχομένου. Και τι γίνεται ακριβώς και με την χρήση των κινηματογραφικών ταινιών στην τηλεόραση. Øh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα και έχω χάσει την αρχή. Είχα την εντύπωση ότι η κυρία Πίτροπος μιλούσε για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχει όμως και μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Στην ε, Σκανδιναβία και ιδίως στη χώρα μου, Δανία, υπάρχει μια υπόθεση με την Apple η οποία έχει μεγάλη ευαισθησία στη χώρα μου, στη Δανία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της κυρίας Επιτρόπου για το πώς πιστεύετε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με μεγάλες πολυεθνικές και πολλές φορές και από τα ίδια τα κάτι μέλη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες ορισμένων εταιριών όταν είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει πρωτοβουλία και παρέμβαση. Τι πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει η Εκτελεστική Επιτροπή, τι προβλέπετε να φέρετε σε νομοθετικό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί ήδη, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη δύσκολο το γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική φορολογία σε επίπεδο ΦΠΑ του των διαφόρων μορφών καλλιτεχνικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Ξέρουμε ότι η χρήση του διαδικτύου για τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει αυξήσει το ΑΕΠ των χωρών μας. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το διαλευκάνουμε. Ο κύριος Τιμπόρκ ήταν φωνή βόντος εν, το, εν τη ερήμο και ζητούσε συνέχεια το θέμα αυτό να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Επομένως σας μεταφέρω και αυτήν την ε, ε αίτησή του. Έρχομαι τώρα σε ένα απονεμένο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι πρέπει να υποστηριχθεί οι, ευρυζωνι, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες αλλά Έχουμε όλοι προβλήματα αυτή τη στιγμή γιατί όλα τα στοιχεία, τα τεχνολογικά τα οποία χρησιμοποιούμε είναι διαφορετικά. Για ένα μικρό επαρχιακό θέατρο, παραδείγματος χάρη, κοστίζει 300.000 η, η χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η σύνδεση με το διαδίκτυο για τα θέματα αυτά. Επόμενο θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προωθήσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά και να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται με καλύτερο τρόπο η αρχιοποίηση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Νομίζω ότι αφήνουμε να χαθεί ένας τεράστιος θησαυρό που είναι οι πρώτες <clears throat> ταινίε του 20ου αιώνα που είναι πολύ δύσκολο πια να ψηφοποιηθούν. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να πάρουμε όλα αυτά τα έργα προτού καταστραφούν τελείως και να τα εκμεταλλευτούμε αλλά το έργο είναι ποιος μπορεί να επιφορτιστεί με το, ε, με το εγχείρημα αυτό. Είναι λοιπόν ένα θησαυρό καλλιτεχνικό όλε αυτέ οι ταινίε αρχέ του 20ου αιώνα που δεν πρέπει να χαθούν. Έχουμε επίση Έχουμε παραγωγή χάρη πίνακες από προηγούμενους αιώνες, τους οποίους διατηρούμε, αλλά δεν διατηρούμε τις ταινίε αυτές από τις αρχές του 20ου αιώνα, που θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διατηρηθούν. 20 λεπτά για να απαντήσετε, κύριε Επίτροπε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσες. Αποτελούν πρόκληση και τόσο για εσάς όσο και για εμάς. Μου έκανε εντύπωση η παρατήρηση της κυρίας Μακλάρκεν ότι μερικές φορές ε, η τεχνολογία πήγαινε με τέτοια ταχύτητα που εμείς συζητάμε νομοθεσία και ξαφνικά έχει ήδη περάσει από μπροστά μας η τεχνολογία συγκεκριμένη θα έλεγα και ένα από τα πράγματα που με κάνει και νιώθω δύσκολα παρότι δεν δυσκολεύουμε ιδιαίτερα στη δουλειά μου. Ποτέ δεν έχω δουλέψει με τόσο ξέφρενους ρυθμούς όσο αυτή τη στιγμή. Εξακολουθώ να απολαμβάνω τη δουλειά μου, οπότε μην ανησυχείτε. Αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο και χρειάζεται πολύ χρόνο η δημοκρατία 27 κρατών μελών και μπορώ να το εξηγήσω στον εξωτερικό κόσμο και με ένα κοινοβούλιο που συμμετέχει πραγματικά και με συναδέλφους που πραγματικά ενδιαφέρονται σε ορισμένα ζητήματα όπου θέλουν να υπάρξουν ευκαιρίες ε, συνολικά όμως ε, είναι χρονοβόρα η διαδικασία και εμείς είμαστε όλο και πιο υπεύθυνοι για να εξηγήσουμε στον εξωτερικό κόσμο ότι μας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα και ότι τα μελετάμε. Για να σας αναφέρω ένα για παράδειγμα. Το αναφέρατε δύο από εσάς, η προστασία των ανηλίκων. Όπως υπόθηκε πολύ σωστά, η εκδήλωση στη Washington θα είχε αποτελέσει μια καταπληκτική ευκαιρία, αλλά δυστυχώς η φύση εκεί μας επιβλήθηκε. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο η Τζάνα υπογράψαμε τη συμφωνία. Αυτό που είναι ακόμα σημαντικότερο από την υπογραφή ενός εγγράφου υποσχεθήκαμε ότι για όσο χρόνο θα παραμείνει σε αυτό το χαρτοφυλάκιο να συνεργαστούμε. Χαίρομαι λοιπόν που εκφράστηκε αυτή η επιθυμία, αλλά είπαμε, είμαι στην άλλη ότι στο τέλος της Άνοιξης καλό θα ήταν να κάνουμε μια συνάντηση, μια, ένα συνέδριο μαζί με τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και τις ΗΠΑ για αυτό το ζήτημα και να εμπλακούμε περισσότερο και να λάβουμε περισσότερε πρακτικέ συμβουλέ, όπω ελπίζουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχω επίση την αίσθηση ότι είναι σημαντικό ζήτημα το δικαίωμα του να σας ξεχάσουν, για παράδειγμα, να μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας στο διαδικτύο, αλλά μην κατηγορείτε τον εξωτερικό κόσμο για λάθη δικά σας. Αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι παρότι υπάρχει ένα πλήκτρο delete μην περιμένετε ότι αυτό σβήνει τα πάντα. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα με το οποίο ασχολούμαι ενεργά. Είναι μια διαδικασία όπου, που αφορά όχι μόνο την επικοινωνία με τα παιδιά, αλλά την επικοινωνία και με γονείς, με δασκάλους, με τους τομείς, με τις βιομηχανίες, αναμφίβολα, αλλά εν τέλει σκοπός μας είναι να προστατέψουμε τους πιο ευάλωτους. Ένα άλλο ζήτημα ειλικρινά αναφέρω ότι αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι στην Επιτροπή σας ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πολιτισμός, τόσοι πολυπολιτισμοί, γλώσσες, τόσες πολλές γλώσσες, η κληρονομιά μας αλλά και η δημοκρατία. Μιλάμε και για δημοκρατία και ότι ακόμα προσπαθούμε να την επιτύχουμε. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό που ανέφερε ο Μάρτιν. Αντιλαμβάνουμε ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια, στο ίδιο στάδιο. Μιλάμε για ελευθερία λόγου και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυμορφία, τον πλουραλισμό την ημέρα των ευχαριστειών Δυσκολεύτηκα να επικοινωνήσω με ανθρώπους από την Apple. Υπάρχει διαφορά ώρας 9 ε, ώρων. Ε, ήταν δύσκολο λοιπόν σήμερα το πρωί να μπορούσα να μιλήσω τηλεφωνικά. Ζητάω διαφάνεια. Δεν μπορώ να αναγκάσω μια επιχείρηση να αλλάξει το επιχειρησιακό τη μοντέλο. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να εξαρτάται από μένα ή από την Κομισιόν. Αλλά αυτό που μπορώ να απαιτήσω είναι να υπάρχει διαφάνεια, να γνωρίζουμε το διακύβευμα και τι πρέπει να προσδοκούμε από τις δραστηριότητε, μια εταιρεία όπω η Apple. Για να σας μιλήσω τώρα για το Connected TV για τη συνδεδεμένη τηλεόραση. Η πράσινη βίβλο θα υιοθετηθεί στις αρχέ του επόμενου έτους. Γι' αυτό λοιπόν ε, επιτρέψτε δύο μήνες ακόμα και μετά θα είναι έτοιμη η πιθανή αναθεώρηση του AVMSD. Δεν μπορώ να προβλέψω που θα καταλήξουν οι δεβουλεύσεις και εκεί συζητάμε. Ακόμα από ότι χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο, κάποιοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να αλλάξουν ορισμένου κανόνε, το γνωρίζουμε. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι πολύ πρώιμη μια αλλαγή του ADMST. Να σας δώσω και εδώ άλλο ένα παράδειγμα που αφορά ολόκληρο το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν μιλάμε για την οδηγία του 2001 μπορεί κάποιος να λέει ότι δεν είναι απόλυτη προτεραιότητα αλλά σήμερα σε αυτό το τομέα οδηγία του 2001 ισχύει ακόμα ενώ υπάρχουν τόσο τεράστιες αλλαγές στον κόσμο. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη όχι τον αριθμό των ετών αλλά την κατάσταση της αγοράς. Το πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Όλους τους παράγοντες τώρα η Συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού, μιλώντα για τη συνδεδεμένη τηλεόραση, είναι πολύ ενδιαφέρον μεταξύ παραδοσιακών εταιριών εκπομπή ε, και νέων. Η AVMST περιλαμβάνει κανόνε για γραμμικέ και μη γραμμικέ ε, υπηρεσίε, κάνει τη διάκριση επιλογή και χρήση. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πώ οι μελλοντικέ εξελίξει μπορεί να αλλάξουν την ισορροπία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που τίθεται και κατά πόσο το παρόν πλαίσιο εξακολουθεί να είναι καλά προσαρμοσμένο στην κατάσταση που Και κάτι τέτοιο. Και αυτό αποτελεί ένα ενδεχόμενο. Ενημερωνόμαστε και θα σα ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Μιλώντα τώρα για την Ουγγαρία, μια από τις ε, δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια τη τη και τη συνάντησή μου με τους ακτιβιστές, ε, δημοσιογράφους, ότι μας εξηγούσαν τι συνέβαινε στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Ένα από κοινά τα ζητήματα που το περίμενα ήταν τι κάνετε εσείς στις δικές σας χώρες και η Ουγγαρία αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Θα ξεκινήσω με μια θετική νότα μιλώντας για την Ουγγαρία ότι κοιτώντα την Ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως προτάθηκε ήδη στην Ουγγαρία οι αλλαγές δεν αντιμετωπίζουν όλα τα εκκρεμόντα ζητήματα που με απασχολούν. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ανησυχίες από πλευράς μου και θέλω η Ουγγαρία να συνεχίσει το διάλογό της με το Συμβούλιο αλλά και να αναλάβει περαιτέρω δράση. Με άλλα λόγια, δεν είναι αρκετό να μας λέει η κυβέρνηση ότι συζητάει με το Συμβούλιο. Πρέπει να δράσει. Κάτι ενδιαφέρον που συνέβη στον Πακού, στο Αζερμπαϊτζάν, σε εκείνη τη συνεδρίαση, με συνόδευε με άλλους δύο επιτρόπους ο Επίτροπος για τον ΩΣΑ και του Συμβουλίου αυτοί μίλησαν πιο ανοιχτά από ότι εγώ. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω πιο διπλωματικά, αλλά ήμουν σαφής, χωρίς κανένα δισταγμό. Ακούγοντας τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, του είπα στο τέλος, Θεέ μου, αν μπορούσες να μιλήσεις ε, στο δικό σου λαό που στην Ουγγαρία θα αισθανόμουν ανακουφισμένοι. Ας περιμένουμε λοιπόν και να δούμε. Θέλω να δω δηλαδή άμεση δράση για αυτό το ζήτημα ώστε πραγματικά να επιτευχθεί πραγματική ανεξαρτησία online όπως και σε άλλες χώρες. Κυρία Κάμερεβερντ, μιλώντας για το Ντουμπάι, είναι συναρπαστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι μια εκδήλωση πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Πάντα είναι ενδιαφέρον βέβαια το θέμα αυτό, αλλά αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον θα έλεγα, διότι αφορά τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες υπό τις σημερινές περιστάσεις. Το περιεχόμενο λοιπόν και όπως πολύ σωστά αναφέρατε ορισμένα μέλη έχουν ήδη ε, πεπεφρασμένες ε, ε, απόψεις και οράματα λυπούμε που ορισμένοι δεν ακούν ο ένας τον άλλο πάντα θέλω εγώ να ακούω και όσους έχουν άλλες ιδέες από μένα ώστε να ακούσω τα επιχειρήματα να τα πάρω και ίσως και να αντικαταστήσω αν χρειάζεται θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ανασκόπηση αυτού του συνεδρίου για να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογή αυτή τη συνθήκη ATR και εμεί θα προσπαθήσουμε να ενταχθούμε σε αυτό το πλαίσιο Κομισιόν Μέχρι στιγμή έχει εκφράσει την υποστήριξή τη και επιφυλάσσει το οποιοδήποτε δικαιώματο αναζήτηση διορθωτικών μέτρων δυνάμεων των συνθήκων και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει την αντιμετώπιση του ζητήματο μια εξαιρετικά καλά ενημερωμένη και ικανή αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι. Τώρα όταν μιλάτε για ορφανά έργα, πολύ σωστά, η οδηγία μπορεί να διευκολύνει την αδειοδότηση για ορισμένα αρχαιοθετημένα έργα και θα βοηθήσει ευκολότερη πρόσβαση online στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε, αν δεν δραστηριοποιηθούμε και αν δεν έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει, χάνουμε χρόνο, θα χάσουμε έναν αιώνα ολόκληρο. έναν αιώνα και τώρα συζητώντας για το Ευρωπαϊκό όταν κάνουμε ένα σωρό πράγματα σωστά αλλά χάνουμε την πτυχή όπου ε, υπάρχουν τόσα πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν αναφέρονται εκεί μέσα, τότε χάνουμε μια ευκαιρία. Η οδηγία λοιπόν είναι ένα στοιχείο για την καθιέρωση της ψηφιακής ενίας αγοράς, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εύκολη πρόσβαση σε όλο το δημιουργικό περιεχόμενο βάσει καινοτόμων και διασυνοριακών επιχειρησιακών μοντέλων. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει στόχος μας. Και μιλώντας για την να ξανά είναι τόσο κοντινή σε μας. Ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Κυρία Κώστα, όσον αφορά την κινηματογραφική κληρονομιά, προετοιμάζουμε μία πρόταση για τον ψηφιακό κινηματογράφο που θα καλύπτει την ε, κινηματογραφική κληρονομιά, την ψηφιοποίηση του κινηματογράφου και σύνδεση online στις αρχές του επόμενου έτους. Δεν απομένει δηλαδή πολύ καιρός. σχετικά με το θέμα του ΦΠΑ, Πρόεδρε. Κατά κάποιο τρόπο, τίθεται εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας. Εάν πράγματι εμείς προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι με τη νέα τεχνολογία δημιουργούνται νέες μορφές παρουσίασης του περιεχομένου, χωρίς να παρουσιάζουμε το περιεχόμενο, αυτό δεν έχει σημασία και δεν θα είμαστε έτσι ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ΦΠΑ. Και αυτό θα είναι κρίμα. Ίσως να είμαι λίγο δυσάρεστη. Όταν σας σκέπτομαι και κάπου κάπου σας σκέπτομαι, σκέπτομαι μικρές αίθουσες κινηματογράφου και θεάτρου, έτσι με έχετε επηρεάσει. Πάντω παρόλα αυτά πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ δεν ξεχνώ αυτά τα οποία μου έχετε ζητήσει και σα στηρίζω σε αυτά που έχετε κάνει γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα για τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες. Αναζητούμε λοιπόν λύσεις. Δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε τις ε, εξελίξεις στον τομέα του φάσματος. Ε, είναι θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί τελικά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες αυτού του κλάδου, αυτού του τομέα. Δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις εκεί όπου μπορούμε και ελπίζω να μπορέσουμε στο τέλος να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανάπτυξη όλα των μέσων και ξέρετε ότι δημιουργούνται όλο και περισσότερα τέτοια μέσα και αυτά θα πρέπει να καλύψουμε στα πλαίσια αυτών που σας απασχολούν. Ευχαριστώ Επίτροπε. Μία επιπλέον ερώτηση. Νομίζω ότι είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Ε, στις Κάνες, στο φεστιβάλ του κινηματογράφου, την παρουσία πολλών σκηνοθετών Είχατε μιλήσει για το Ausweitungsfenster. Το παράθυρο διεύρυνσης κατά κάποιο τρόπο. Όταν έχετε μια ταινία στι ε, στις οθόνες υπάρχει ένας χρόνος ε, προτού μπορέσει να κυκλοφορήσει σε άλλο φόρμα, όπως παραδείγματο χάρη υπομορφή DVD. Και η Κομισιόν, από ό,τι βλέπω, θέλει να μικρύνει αυτό το παράθυρο, την απόσταση κατά κάποιο τρόπο, τη χρονική απόσταση γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνει κανείς στο σινεμά και να βλέπει ένα έργο. Θα τα παίρνει όλα σε DVD, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και οι αντίπαλοι που λένε ότι θέλουν να έχουν μόλις δουν το έργο και το DVD. Είναι λοιπόν ένα σφάλμα η στάση της Κομισιόν ή θα μπορούσε να την δικαιολογήσει και να επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτής της πρότασης Κομισιόν. Είμαι μέλος της Κομισιόν, οπότε μπορείτε να θέτετε όλες τις ερωτήσεις. Και αν δεν μπορώ εγώ να απαντήσω, θα αντιθέσω στους συναδέλφους μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, δεν ήταν ποιο είχα πει. Πράγματι εδώ τίθεται το θέμα της στενής συνεργασίας με την ε, Επίτροπο ε, Βασιλείου. Σκύλα από τη μία χάρη από την άλλη. Να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα τι εννοώ. Το θέμα είναι να πάρουμε μέτρα τα οποία δεν θα λειτουργήσουν ε, αρνητικά για τον κινηματογράφο. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό. Οι αριθμοί πάντως δεν δείχνουν να υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος και θα πρέπει αυτοί που εμπλέκονται εμπορικά στην παραγωγή ταινιών να ε, ξεκαθαρίσουν τις επιλογές τους. το να είναι δυνατόν να κατεβάσει κανείς τα έργα αυτά νωρίτερα, αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζει, θα έλεγα, και τις αντιδράσεις του κόσμου. Και μένουμε και στα πλαίσια του νόμιμου, αν θέλετε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα παράνομης ε, γενικά χρήσης του υλικού αυτού Ξέρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, σαν παράδειγμα, τα παιδιά στην Ολλανδία. Είχα πάει σε ένα σχολείο και ένας 14χρονο, ο οποίος μου είπε, κοιτάξτε, ό,τι θέλετε μπορώ να σα το κατεβάσω εγώ ή αν δεν θέλετε να σας μάθω εγώ πώς να το κατεβάζετε. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση υπάρχει. Ο κόσμος εν τω μεταξύ έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, οι νέοι, αλλά όχι μόνο οι νέοι και είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων Το θέμα δεν είναι αν νομίζω εγώ ότι κάτι τέτοιο έχει νόημα, αλλά αν πράγματι έχει νόημα. Και να μην μπούμε σε αυτή τη φάση στη συζήτηση για το ελεύθερο διαδίκτυο το οποίο είχατε θέσει, γιατί εκεί πράγματι θα υπάρξουν πάρα πολλές παρανοήσεις. Καταλαβαίνετε ε, τι εννοώ με αυτό. Ελεύθερο ίντερνετ αλλά με κανόνες παιχνιδιών. Καλώς λέει η Πρόεδρος, θα κλείσει εδώ η συζήτηση. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Χαιρετισμού στους Υπουργούς Πολιτισμού. Πρέπει να μας βοηθήσουν να τους πείτε για να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά εκεί όπου εμείς επιθυμούμε. Σημείο 4 τώρα της ημερησίας διάταξης. Παραμένουμε στον ίδιο συνδεδεμένο κόσμο. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Κάμερε Φέρτ, η οποία έχει προετοιμάσει και την ομιλία της με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει και το μικρόφωνο της ε, η κυρία Κάμερα Φέρτ. Αυτό είναι πρώτα μια, ένα αδρό γράφημα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω μια πλήρη εισαγωγή σε όλα τα θέματα της ε, συνδεδεμένης τηλεόρασης, γιατί ίσως κάποια άλλη φορά θα μπορέσω να το κάνω πιο απτό. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι η τεχνολογία κάνει δυνατό τα προγράμματα του ραδιοφώνου και του ίντερνετ και της τηλεόρασης να εμφανίζονται στην ίδια οθόνη της της τηλεόρασης. Αρκεί να έχει η, η οθόνη πέρα της ε, λήψης της τηλεοπτικής να έχει παραγωγικά και μια σύνδεση για το ίντερνετ που μπορεί να το κάνει με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι μπορούν τα κλασικά γραμμικά μέσα όπως είναι η τηλεόραση, να βρίσκονται στην ίδια οθόνη με μη γραμμικά μέσα όπως είναι το διαδίκτυο. Μπορεί κανείς να έχει επαφή με το Facebook ή με άλλα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης μέσα από την ίδια τηλεπτική οθόνη. Δεν ξέρω αν μπορώ τώρα όλα αυτά να σας τα πω. Πρέπει να τα δει κανείς αυτά στην πραγματικότητα το, αυτό το οποίο <clears throat> βλέπουμε είναι ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον για συσκευέ οι οποίε έχουν πολυμορφικό χαρακτήρα. 55% των Βρετανών ήδη έχουν την ε, δυνατότητα να συνδέσουν τη τηλεόρασή του με το ίντερνετ. Μόνο 20% το κάνουν τώρα, αλλά και πολλοί 11% έχουν την πρόθεση να το πράξουν αυτό μέσα στο επόμενο έτος να αγοράσουν μια τηλεόραση Connected TV. Στη Γερμανία προβλέπεται από το Φεβρουάριο του 2013, τουλάχιστον στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις που έχουν ε, επίγεια ψηφιακή τηλεόραση να ανοίξει ένα, μια, δικτυακή πύλη υβριδικής τηλεόρασης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί κανείς να έχει ε, τηλεοπτικές ροές από ψηφιακά μέσα όπως είναι το Spiegel TV, η Web TV κτλ. Ήδη υπάρχουν 13 εκατομμύρια άτομα που έχουν αγοράσει συσκευές Connected TV και το 2003 σε ένα χρόνο υπολογίζεται ότι θα έχουν ξεπεράσει ήδη τα 16 εκατομμύρια και η Samsung είπε το Οκτώβριο του 2012 ότι το προϊόν της, η Smart TV, ήδη έχει δημιουργήσει 10 εκατομμύρια εφαρμογές για, την, ε, για τους χρήστες της τηλεόρασης Connected TV. Επομένως μπορείτε να φανταστείτε ότι στο μέλλον η τηλεόραση που θα έχετε ενώπιόν σας θα μοιάζει περισσότερο με την επιφάνεια χρήστη ενός ε, smartphone ή ενός tablet ε, υπολογιστή. Θα είναι γεμάτη με μικρές εφαρμογές και αυτό φυσικά θα έχει και συνέπειες για όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα νέο βήμα στην σύγκληση των ψηφιακών μέσων και δεν πιστεύω ότι η ρύθμιση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι επαρκής για να προπαρακολουθήσει όλα αυτά τα στοιχεία ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, βιομηχανία τερματικών συσκευών που αποκτά όπως καταλαβαίνετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και η οποία εργάζεται πειρατοδός για να μπορέσει να δώσει στον χρήστη ένα, μια επιφάνεια διαδραστική η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλής ποιότητος αλλά θα διατηρεί και την διαδραστικότητα. Αυτό μας συναρπάζει αλλά ως πολιτικούς για τα μέσα ενημέρωσης μας θέτει ενώπιον ενό καθήκοντο να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για τα νέα αυτά συστήματα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει θεμητός ανταγωνισμός και να υπάρξει και η απαραίτητη προστασία και να εξασφαλίσουμε ότι η κατεύθυνση μετεξέλιξη όλων αυτών των προϊόντων θα τηρεί όλους τους κανόνες του δικαίου καταναλωτών, του δικαιώματο των πνευματικών δημιουργών, του δικαίου ανταγωνισμού κτλ. Όταν λοιπόν μιλάμε για κανονισμούς, μιλάμε όχι μονάχα για τις ε, αρμοδιότητες οι οποίες εμπίπτουν στο έργο της δικής μας Επιτροπής, αλλά είναι και θέματα τα οποία θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες επιτροπές, παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για προστασία καταναλωτών ή προστασία προσωπικών δικαιωμάτων. Στο μέλλον με την Connected TV θα μπορεί κανείς να βλέπει τέσσερις διαφορετικές μορφές μέσων ψηφιακών στην ε, Connected TV. Και γι' αυτό σας έφερα αυτά τα, αυτή την οθόνη την οποία βλέπετε εδώ για να κάνω πιο διαισθητικά ορατή την νέα αυτή πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα πείραμα το οποίο διαμόρφωσε ο κύριος Κόγκλερ, ο του τμήματος μέσων ε, οπτικοακουστικών στο γραφείο του Πρωθυπουργού της Αυστρίας. Έχουμε μια τηλεόραση η οποία έχει σπάσει σε τέσσερα κομμάτια. Πάνω αριστερά βλέπουμε το Χάρι Πότερ. Είναι μια, μια φυσιολογική παρουσίαση μια ταινία. Είναι γραμμικά μέσα. Έχουμε ένα έργο το οποίο ξεκινάει στις 8 η ώρα παραδείγματος χάρη και τελειώνει στις 10 πάνω δεξιά είναι ο Harry Potter επιζητήσει, video on demand. Γιατί μάλλον δεν πρόλαβα να δω το Harry Potter στο έργο και στο μέλλον θα θέλω να τον βλέπω κάποια στιγμή που να έχω εγώ ελεύθερο χρόνο για να μπορέσω να το δω στην τηλεόρασή μου. Αριστερά κάτω έχετε μια ιστοσελίδα από το ίντερνετ. Δηλαδή μπορώ συγχρόνως να κοιτάζω και μια ιστοσελίδα που μιλάει για το Harry Potter, για τη δημιουργία αυτού του έργου, για κομμάτια αυτού του έργου, για τους τοπιούς του έργου, για τα τρίκτα τεχνικά του έργου κτλ. Και στα δεξιά συνεχίζουμε να είμαστε συνδεδεμένοι σε ένα κλασικό ε, teletext, γιατί θέλουμε να παρακολουθήσουμε τι έκανε η Chelsea ή η Arsenal την ίδια στιγμή. Κάθε μία από αυτές τις ε, προσφορές περιεχομένου βρίσκεται και σε ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Είναι χωριστοί αυτοί οι χώροι που αφορούν τη ρύθμιση του καθενό. Σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, το Harry Potter το έργο αυτό, βάσει της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά, θεωρείται ότι ο καταναλωτής είναι απλώς ένας παθητικός αποδέκτης. Και γι' αυτό, σε αυτό το τομέα έχουμε πάρα πολλές ρυθμιστικές διατάξεις. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για αυτούς που έχουν ε, προβλήματα ακοής, πρέπει να μην υπάρχει ε, προτροπή σε πράξεις μίσου, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα ανασκεύαση μιας δήλωσης κτλ. Και θα πρέπει να χωρίζεται η διαφήμιση από το πρόγραμμα. Αν περάσουμε πάνω δεξιά, στο Harry Potter που έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ με video on demand. Δεν είμαστε πια ένας παθητικός καταναλωτής, αλλά ξαφνικά είμαστε ενήλικες καταναλωτές. Γιατί Έχουμε εδώ πέρα ένα μη γραμμικό σήμα στο οποίο μπορούμε εμείς να το κατευθύνουμε με το δικό μας τρόπο. Δεν είναι πια γραμμικό το σήμα. Εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετικές οι προδιαγραφές. Είναι πολύ πιο περιορισμένοι οι περιορισμοί που ισχύουν. Δεν υπάρχει κάποια προδιαγραφή για να διαχωρίζεται η τηλεόραση από το έργο από τη διαφήμιση. Μπορεί κανείς να διαφημίζει παραδείγματος χάρη αλκοολικά προϊόντα, δεν υπάρχει το δικαίωμα να ανασκευάζονται οι δηλώσεις που είναι στο έργο αυτό αλλά φυσικά μπορείτε να δείτε το έργο αυτό όπως θα το βλέπατε και στη τηλεόραση στην ίδια ποιότητα. Αν θέλω τώρα και πάω κάτω αριστερά να βρω περαιτέρω πληροφορίες, πληροφορίες στην ε, οθόνη, βγαίνω τελείω πια από το χώρο της τηλεόρασης και μπαίνω πια στο χώρο του ίντερνετ και στο χώρο εφαρμογής του, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επειδή έχει μονάχα κάποια στοιχεία οπτικοακουστικά. Αυτό, αυτή η ιστοσελίδα που είναι κάποια τρέιλες ή κάποια διαφημιστικά, αλλά γενικά καλύπτεται ως ένα τμήμα του, διαδικτύου. Δεν θα ήταν διανοητό μέσα στην ταινία στο Harry ξαφνικά να βλέπετε ένα σποντ ένα σποτ διαφημιστικό και να έχετε τα πιτσιρίκια να πίνουν σφινάκια, αλκοολικά παραδείγματος χάρη. Αλλά κάτω θα μπορούσε να γίνεται αυτό. Κάτω αριστερά Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο μέσα στο τμήμα πληροφόρηση στο ίντερνετ. Δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμία τέτοια ρύθμιση που να το εμποδίζει. Πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει sponsoring, χορηγία για τι ειδήσει στην τηλεόραση ή ακόμα και στο βίντεο on demand. Στο ίντερνετ όμω ο καθένα μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι sponsor οποιασδήποτε μορφή πληροφορία. Και πάλι μπορεί κανείς να προσθέτει βίντεο, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, όσο εδώ θεωρείται ότι είναι κυρίως ε, περιεχόμενο κειμένου, όλα αυτά μπορούν να προσθεθούν ακόπως και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και κάτω δεξιά στο teletext που βλέπετε, εδώ έχετε πληροφορίες οι οποίες δεν συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επομένως δεν υφίσταται καμία σχεδόν ρύθμιση. Και σε πολλές χώρες όπως τη Γερμανία και η, Αυστρία θεωρείται σαν ένα είδος ραδιοφώνου το teletext. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τέσσερις αυτές περιοχές στην οθόνη σας υπόκειται σε διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες από διαφορετικά μέσα, με διαφορετικούς τρόπους στο σπίτι μας και μέσα από διαφορετικές συσκευές. Οπότε μπορούμε να διαχωρίσουμε την, τα γραμμικά μέσα από τα μη γραμμικά μέσα. Αλλά σε λίγο αυτό δεν θα είναι δυνατό γιατί με την εξέλιξη της τεχνικής όπως βλέπουμε μέσα από την Connected TV αυτή η μορφή διαχωρισμού σε γραμμικά ή μη γραμμικά μέσα δεν θα είναι εφικτή γιατί εμείς ως ε, τηλεθεατές και χρήστες πληροφοριών στο, στο διαδίκτυο θα έχουμε στην ίδια οθόνη και γραμμικά και μη γραμμικά ε, στοιχεία και δεν θα ξέρουμε καν αν βρισκόμαστε στο γραμμικό ή στο μη γραμμικό χώρο των μέσων αυτών. Επομένως εδώ υπάρχει το κίνδυνος ότι η μικρότερη ρύθμιση που υπάρχει στο ένα τμήμα και η μεγαλύτερη ρύθμιση στο άλλο τμήμα θα οδηγήσουν σε μια στρέβλωση ε, ανταγωνισμού. Αν έχουμε μια τηλεόραση ας πούμε, η οποία είναι ιδιωτική, υπόκειται σε ορισμένους κανόνες αλλά χρειάζεται να χρησιμοποιήσει αυτούς τους κανόνες για να ε, δείξουν διαφημίσεις από τις οποίες παίρνουν το κέρδος τους. Ενώ ένα, ένας άλλος πάροχος, ο οποίος είναι ένα είδος διαδικτυακή, δεν υπόκειται για τις διαφημίσεις του στους ίδιους περιορισμούς. Εδώ έχουμε μια στρέβλωση ανταγωνισμού λοιπόν μεταξύ ενός παρόχου κλασικής γραμμικής τηλεόρασης και ενός παρόχου τηλεόρασης επί τη ζητήση. Πρέπει να βρούμε μια λύση για τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν τροποποιήσεις στους κανονισμούς που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τα θέματα αυτά. Και βλέπουμε επίσης ότι μπορεί κανείς να συνδυάσει με όποιο τρόπο θέλει τα, τις διάφορες μορφές περιεχομένου και μπορεί να θέτει στο προσκήνιο ή όχι ένα από αυτά τα τμήματα του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πεπαλαιωμένα τα στοιχεία της ρύθμισης τα οποία υπάρχουν, παραδείγματος χάρη προστασία των νέων, η απαγόρευση των διακρίσεων, η μη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κλπ. Όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωριστούν. Το ερώτημα είναι σε ποιες περιπτώσεις και βάσει ποιων ε, προϋποθέσεων θα πρέπει να εφαρμόσονται όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ισότητα ευκαιριών και ανταγωνισμού και όχι διάκριση. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσει να συνδυαστεί η ρύθμιση όλων αυτών των μορφών περιεχομένου. Αυτό το πείραμα σκέψης το οποίο προσπάθησα να χρησιμοποιήσω για να σας δείξω τη μορφή του προβλήματος δείχνει ότι όλο και περισσότερο με τη σύγκληση των μορφών περιεχομένου κάνει όλο και πιο δύσκολο να υπάρχουν άκαμπτες μορφές ρύθμισης. Μια αντιμετώπιση κατά την άποψή μου θα ήταν στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα να προχωρήσουμε σε μια πιο σαφή ρύθμιση για τους παρόχους πλατφορμών μέσων ε, τη, τηλεόρασης ή διαδικτυακών. Με τον τρόπο αυτό, παραγωγός μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τη διατήρηση του χώρου του ιδιαίτερου που έχει το ραδιόφωνο ή η κλασική τηλεόραση. Μπορούμε να διατηρήσουμε έτσι τη δυνατότητα να κρατήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν για την κοινωνία μας και την ελεύθερη έκφραση η, τηλεόραση και το, η κλασική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή είναι οι τομείς οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τους μεγαλύτερους κανόνες για το, τη μορφή περιεχομένου που θα πρέπει να έχουν και υφίστανται στην μεγαλύτερη ρύθμιση. Το θέμα όμως είναι πώς μπορούμε αυτά τα ε, πλεονεκτήματα που φέρει η μορφή αυτή που έχουν να διατηρηθούν και στη νέα μορφή Connected TV. Αν εμείς μπορούμε να σκεφτούμε μια οθόνη όπου τρέχουν διάφορες εφαρμογές συγχρόνως, το ερώτημα είναι πού θα μπορεί να βρει κανείς το κλασικό ραδιόφωνο ή την κλαστική τηλεόραση. Στην πρώτη σελίδα βλέπω τα επίσημα τα κρατικά προγράμματα τηλεόραση ραδιοφώνου στην πρώτη σελίδα ή στην τελευταία σελίδα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι προσβάσιμο ή θα τα βρω μονάχα στο τέλος ενώ στην πρώτη σελίδα θα έχω το Apple TV, θα έχω το Facebook ή αυτά τα οποία έχει προτείνει ο κατασκευαστής της συσκευής. Επομένως, τίθεται το ερώτημα αν μπορώ να βρω μια λύση ώστε η προνομιακή μεταχείριση να συνδέεται με μεγαλύτερη ρύθμιση, με περισσότερους κανόνες και να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ προνομιακής μεταχείρισης και ρύθμισης. Και όπως σας είπα προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του κατασκευαστή αυτών των συσκευών, γιατί στο μέλλον ο κατασκευαστής ήδη θα ξέρει πώς θα είναι η οθόνη στο μέλλον. Αυτός ξέρει πώς θα είναι η οθόνη που θα δω εγώ πρώτη φορά όταν τη βάλω στην πρίζα. Θα ξέρει ήδη ποια είναι τα πράγματα τα οποία προκρίνονται πρώτα, τα οποία φαίνονται πρώτα στον ε, χρήστη. Θα είναι τα κλασικά προγράμματα τηλεόρασης ή θα είναι κάτι άλλο. Και πώς τα συνδέει αυτά μεταξύ τους ο κατασκευαστής. Υπάρχει εδώ κάποια υποχρέωση λοιπόν για τον κατασκευαστή ότι κάποιες ε, μορφές περιεχομένου που έχουν μεγαλύτερη ρυθμιστική πυκνότητα και ε, βάρος θα πρέπει να τίθενται σε πιο περίοπτες θέσεις. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της δυνατότητα ανώνυμης χρήσης της τηλεόρασης. Και εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε κανόνες που επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει τη τηλεόρασή του παραμένοντας ανώνυμος. Το να έχουμε τώρα, όπως παραγωγός χάρη στην υβριδική τηλεόραση, μια αξιοποίηση του θεατή και με τον τρόπο αυτό μπορεί φυσικά ο κατασκευαστής να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο το καταναλωτή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαγορευτεί κατά τη δική μου απόψη και αυτό έχει νόημα μονάχα να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τα προβλήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό αφορά φυσικά και την εξέλιξη των ίδιων των συσκευών που θα πρέπει να έχουν τη λεγόμενη ιδιωτικότητα εξ αρχής, δηλαδή η κατασκευή τους να είναι τέτοια, ώστε να προστατεύει την ιδιωτικότητα του χρηστή και να μην αποκαλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία. Και επομένως μέσα στα πρότυπα τα οποία προβλέπονται, πιστεύω ότι θα πρέπει πάντα να υπάρχει δυνατότητα, εάν εγώ σαν χρήστης δεν πω κάτι διαφορετικό, να προστατεύω τα δεδομένα μου. Μια προσωπικοποίηση αυτής της ε, οθόνης λοιπόν και της επιφάνειας επαφής θα πρέπει να γίνεται μονάχα με την πρωτοβουλία του χρήστη. Ως ε, χρήστης λοιπόν της Connected TV, ως ε, θεατής της τηλεόρασης θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα εγώ να αποφασίσω με το δικό μου τρόπο τι θέλω να βλέπω και τι είδους πληροφορίες θέλω να πάρω από τον πάροχο υπηρεσιών ή από τον κατασκευαστή. Επίση, προστασία των νέων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά φυσικά μόνο το διαδίκτυο, αλλά θα αφορά και την υβριδική ή συνδεδεμένη τηλεόραση και θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το θέμα αυτό. Αυτό, όπως ξέρετε, μέχρι στιγμής έχει εθνικό χαρακτήρα το δίκαιο προστασίας των ε, νέων. Έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα όταν πρόκειται για το ποιε πρέπει να είναι οι, οι ε, εκπομπές που δεν θα πρέπει να διακόπτουν από διαφημιστικά σπότ όπως είναι οι παιδικές εκπομπές ή ποιες εκπομπές δεν θα πρέπει να προβάλλονται όταν ε, είναι ώρες που είναι στην τηλεόραση οι νέοι κτλ. Αλλά υπάρχει και το ερώτημα του κατά πόσο στο μέλλον θα είναι δυνατόν να έχουμε κατασταλτικά μέτρα προστασίας των νέων και αν θα είναι εφικτό να εφαρμόσονται. Στη Γερμανία τους προηγούμενους μήνες είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα αυτά η, τα κρατήδια στη Γερμανία ήδη έχουν ε, διαφορετικές απόψεις πολλές φορές και δεν έχουν πείσει ορισμένα ότι πρέπει να υπάρχει μια κατασταλτική αντιμετώπιση. Επομένως θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς την προληπτική ρύθμιση για τα θέματα αυτά και αυτό αφορά και μια συνολική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα-δύο σημεία μόνο ακόμα θέλω να αναφέρω. Το θέμα της Connected TV και του τρόπου με τον οποίο θα κάνουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις είναι σαφές ότι δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό η έκθεση που εγώ θέλω να παρουσιάσω δεν θα κομίσει μια συνολική λύση για όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε να θέσουμε κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις επί των οποίων η Κομισιόν θα κάνει μια περαιτέρω επεξεργασία και ότι με τον δικό μας τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε μερικά σημεία για το τι πρέπει να περιέχεται στο περιεχόμενο της ε, τηλεόρασης, ποια θα είναι τα ελάχιστα ε, κανάλια ή υπηρεσίες που θα πρέπει να περιέχουν, πώς θα εξασφαλιστεί η ακαιρεότητα των ε, εκπομπών και όχι να τίθεται πάνω τους μια διαφήμιση ανα πάσα στιγμή να διακόπτονται από, τη, από διαφημιστικά σποτ. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν της ακαιρεότητας του τηλεοπτικού σήματος και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να επιτρέπει είτε ο ίδιος ο χρήστης επιτρέπει να έχουν αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες, τα overlays όπως λέγονται και ποτέ δεν θέλει να τα έχει και επίσης ο αυτός ο οποίος εκπέμπει να έχει έναν τρόπο να αποτρέψει άλλους από το να θέτουν διαφημίσεις πάνω στο δικό του περιεχόμενο. Δεν μπορεί λοιπόν τη στιγμή που δείχνει ένα κανάλι τα νέα της ημέρας κάποιος άλλος να προσθέτει σε αυτό διαφημίσεις. Το ερώτημα είναι λοιπόν επίσης πώς μπορούμε να αφήσουμε συστήματα τα οποία είναι κλειστά είναι προπριετέροι ή αν θα έχουμε λύσεις που θα επιβάλλουν σε όλους να έχουν ένα ελάχιστο περιεχόμενο και αν είναι συστήματα κλειστά να εξασφαλίζουμε ότι δίνουν κάποια πρόσβαση στα, στις βασικές υπηρεσίες. Είναι κάπως δύσκολο να αποφύγει κανείς τις προσπάθειες να δώσει κανείς μια λύση πακέτο, εξού και ένα κλειστό σύστημα και να θεωρεί κανείς ότι μπορεί ο κατασκευαστής να πει καταναλωτή ξέρω ότι θέλεις και στα δίνω. Σου δίνω ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεσαι και τίποτα παραπάνω. Αυτά είναι τα κλειστά συστήματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μην περιορίσουμε τη δυνατότητα λήψης απόφασης του καταναλωτή και να διατηρήσουμε συγχρόνως την πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης. Και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να εξασφαλίσει την πολυμορφία των μέσων, την ισότητα ανταγωνισμού, την δυνατότητα ευρείας πρόσβασης και την προστασία των ασθενεστέρων χρηστών, όλα αυτά απαιτούν μια κοινή συνένεση, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά βρίσκονται στη βάση της ε, δημοκρατίας μας και είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές μέσα σε οποιαδήποτε ρύθμιση η οποία θα γίνει για τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά άπτονται άμεσα της δημοκρατίας μας και είναι βασικά στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας και γι' αυτό θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην γίνει με αυτές τις προηγούμενες ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και οι οποίες εμπόδισαν την πραγματική ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστω θα σας χειροκροτούσα, λέει η κυρία Πακ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και η προβληματική που μας παρουσιάσατε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ο Ζαν Μαρίτα θυμάται αυτά και η Πέτρα επίσης όταν είχαμε αντιμετωπίσει την οδηγία, τη δεύτερη οδηγία για την τηλεόραση. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσουμε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι περίπου ο τετραγωνισμός του κύκλου. Αλλά σου είμαι πάρα πολύ ε, ευγνώμων, Πέτρα, μου έχεις ανοίξει τα μάτια για πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω τώρα τι είναι ε, εφικτό ή όχι, αλλά εγώ προσωπικά θέλω να μπορώ να βλέπω την τηλεόραση όπως έχω κάνει μέχρι τώρα, χωρίς να με πίζουν στην προπαγάνδα και δεν θέλω να έχω διαφημίσεις από τη μια μεριά και από την άλλη κάθε 10 ή 20 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία λες θα πρέπει να είναι εφικτά. Περιμένουμε τώρα το έγγραφο εργασία σου το Φεβρουάριο, αλλά περιμένουμε και από την Κομισιόν να αντιδράσει. Μπαίνουμε σε ένα νέο χώρο τελείω, όλα αυτά είναι φυσιολογικά, είναι απείρως ταχύτερη τεχνολογία από ότι η πολιτική. Ήδη όπως ακούσαμε και από την Έλλη Κρούς. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω τα λόγια στον Ζωάν Μαρή Καβαντά, ο οποίος είναι γνώστης και μύστης των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάμερβερτ, την κυρία Πρόεδρε, τον ειδικό. Ευχαριστούμε την κυρία Κάμερβερτ γιατί ασχολήθηκε και ανέλησε πολύ θεμελιώδη και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Για να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση, την περασμένη εβδομάδα πέρασα μια ημέρα σε έναν φορέα τηλεοπτικών εκπομπών με το συνδυασμό των διαφορών box από τον Google μέχρι άλλα που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε διάφορα πράγματα στις οθόνες μας. Έχετε πολλά ερωτήματα όπου πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα προφύλαξης αλλά και κίνητρα. Θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά Αυτό που μας μένει από την έκθεσή σας ουσιαστικά και από την πραγματικότητα όταν βλέπουμε γιατί πρόκειται και πώς λειτουργεί είναι ότι πρώτα απ' όλα για κάποιο καιρό ακόμα, αρκετό καιρό ακόμα η τηλεόραση γύρω από την οποία καθόμαστε θα αποτελεί το βασικό μέσο η εκπομπή, η μετάδοση των προγραμμάτων και οι τηλεθέτες ε, αλλά Επιχειρούνται αυτή τη στιγμή διάφορες άλλες τεχνικές και καλό θα ήταν να προβληματιστούμε πραγματικά για το πώς ε, θα ελέγξουμε αυτή την υπόθεση έτσι ώστε να είναι ωφέλιμη για τους τηλεθεατές. Υπενθυμίζω ότι οι τηλεθεατές με το Connected TV ουσιαστικά ο τηλεθεατής κατευθύνει τα δικά του προγράμματα τα οποία προβάλλει το Connected TV τα οποία μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε στον κόσμο Εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που αναφέρατε, τις εξαιρέσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά των online οπτικοακουστικών ε, υπηρεσιών βασίζεται σε διαφορετικούς αισθητά οικονομικούς μηχανισμούς ε, από ό,τι στα κλασικά οπτικά ακουστικά μέσα, RGNA ή ψηφιακά τις κλασικές ουσιαστικά θα λέγαμε τηλεόραση πρόσβαση στο περιεχόμενο στο διαδίκτυο αποτελεί τεράστια πρόοδο για τους τηλεθεατές καθώς και για τους χρήστες του διαδικτύου Ουσιαστικά υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες επιλογής. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και παγίδα. Εξάλλου αυτό αποτελεί ευκαιρία για τους Ευρωπαίους φορείς την την ε, ελεγκτές ε, διανομής προγραμμάτων να αξιοποιήσουν το πολιτιστικό μας ε, πλούτο σε παγκόσμιο επίπεδο και να βρουν ε, καινοτόμους τρόπους κατανάλωσης που θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εξακολουθεί να αληθεύει ότι η εμφάνιση της ε, Connected TV που θα ανατρέψει το οπτικό ακουστικό τοπίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε καλύτερη άρθρωση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών με τα μέσα ρύθμισης που υπάρχουν ήδη αφετέρου σε ευρωπαϊκό, ε, σε ευρωπαϊκό και αφετέρου σε διεθνές επίπεδο. Η εξέλιξη τώρα του Connected TV όσον αφορά την ανταλλαγή αγαθών και τις αμοιβέ των δημιουργών θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο συζητήσεων εμπεριστατωμένων όχι μόνο όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών του περιεχομένου και της αμοιβή των μηχανισμών αναζήτησης αλλά και στα προγράμματα που θα εκπέπονται. Θα πρέπει δηλαδή να επαναπρογραμματιστούμε όσον αφορά το όλο ζήτημα δεδομένων των τεχνολογικών εξελίσεων και των αγορών που υλοποιούνται. Για να μην γίνει η συνδεδεμένη τηλεόραση μια ζούγκλα, σκοπιμό θα ήταν στο σχέδιο έκθεσης ε, να αναφέρεται η ευθύνη των εκδοτών, να ορίζεται ο ρόλος του παρόχου υπηρεσιών πολυμέσων και η έννοια του προγράμματος που θα χρήζει δυναμική ερμηνεία που να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της ε, ε, εκπομπής, ε, τηλεοπτικών εκπομπών δεδομένων των εκτιμάτων 24 και 25 της οδηγίας για τα οπτικά ακουστικά μέσα Αφετέρου, δεδομένου του ανταγωνισμού πολλών κυρίως αμερικανικών εταιριών που έχουν προοδεύσει ιδιαίτερα και προαρέχουν από κακουστική υπηρεσία αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καινοτόμε προσφορές. Και γνωρίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είμαστε, έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, θα πρέπει να σκεφτούμε την προσαρμογή των κατάλληλων αγορών στις εξελίξεις ε, του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού κόσμου με δυναμικό τρόπο ώστε να διατηρηθεί ο δημιουργικός ανεξάρτητος ιστός τον οποίο χρειαζόμαστε απολύτως. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με τις περισσότερες από τις συστάσεις σας, αγαπητή κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ, Ζαμάρη. Κυρία Έμα Μακλάρκιν. Thank you. Ευχαριστώ. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στην Επιτροπή αυτή τις ευκαιρίες που μας ανοίγει το διαδίκτυο και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο μέσω της λεγόμενης connected τηλεόρασης. Το θέμα είναι ότι όπως είπατε θα πρέπει να προλαμβάνουμε όλες, να, ναι ακριβώς να συμβαδίζουμε με όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και αυτά τα τεράστια βήματα σχετικά με το μέγεθος αυτό το οποίο είπατε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες στη χρήση της εικόνας της τηλεόρασης και παρέμβαση στην εικόνα της τηλεόρασης. Απαραίτητο βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα είναι το, ε, η υψηλή ταχύτητα, εν γιατί σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο δεν είναι παντού εφικτό. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τον τρόπο λειτουργίας της διαφήμισης στα πλαίσια αυτής της νέου τύπου τηλεόρασης. Η διαδικασία τώρα ξεκινάει και αυτό είναι καλό γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιο χρόνο για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε γιατί ανησυχώ λίγο ότι όλα αυτά τα μέσα είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους και διαρωτώ σε ποιο βαθμό λεπτομέρειας μπορούμε να φτάσουμε στα πλαίσια της ρύθμισης. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές λοιπόν και σε αυτή τη φάση θα εξαρτηθεί από μας το πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ Πέτρα για την επισκόπηση που μας έδωσε. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικός αυτός ο χώρος και θα πρέπει να συζητήσουμε σίγουρα περισσότερο για τα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες στο θέμα της Connected TV από ό,τι είχαμε σκεφτεί στην αρχή. Πολύ περισσότερο από ότι με τις συσκευέ που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, αν μπορούμε όλα αυτά τα, τις ροές περιεχομένου να τις ε, συνδυάσουμε σε μία επιφάνεια μονάχα, αυτό δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητε στο χρήστη. Μπορεί να προσθέσει και ένα ακόμα μέσο. Να έχουμε παραγωγή τα έντυπα μέσια. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί να συνδέσει με ένα κτυπωτή παραγωγός χάρη την τηλεόραση. Και πάλι είναι το θέμα της πρόσβασης σε όλα αυτά τα θέματα. Το βασικό ερώτημα όμως είναι πώς μπορώ εγώ σαν χρήστης να έχω πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και πώς μπορεί να είναι ενεργός ο χρήστης και πώς να μπορεί να επιλέγει τις διάφορες μορφές διαφημίσεις οι οποίες πολλές φορές υποβολημία θα παρουσιάζονται. Να υπάρχει δυνατότητα της επιλογής λοιπόν. Και όπως είπες υπάρχει και η ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και μια δυνατότητα ανωνυμοποιημένης πρόσβασης και ουδετερότητος όταν κανείς χρησιμοποιεί αυτούς τις νέες μορφές τηλεόρασης. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα είναι πώς να μπορέσει κανείς να περάσει σε ορισμένε μορφές περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται να περάσει από τις, ε, από τις κλίδες που θέτει κάποιος άλλος και δεύτερον πώς θα εξασφαλίσουμε την ισότητα α, ε, ανταγωνισμού. και να εξασφαλίσουμε φυσικά και ότι θα διατηρήσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν οι υπηρεσίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα αναδυθούν. Η Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία Λορένα Αλόνσο. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ εκτιμάμε ιδιαίτερα αυτή την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μας. Τα όσα ακούσαμε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε αναγνωρίσει, κυρία Κάμερμπερκ, πολλά από τα ζητήματα που βρίσκονται όντως στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, όπως αναφέρατε και όπως αναφέραν και ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Τώρα ξεκινάει αυτό το στάδιο της σύγκλησης και στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι ακριβώς να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ώστε καθώς προχωράει γρήγορα η τεχνολογία να έχουμε ξεκινήσει αρκετά νωρίς να συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Και στη συνέχεια θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματο. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις, λεπτομέρειες, αντιδράσεις. Ευχαριστώ αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ για σήμερα. Έχουμε πάρει. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Στην εισηγήτρια δίνω το λόγο λοιπόν για τέλος. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα αντιμετωπίσουμε και στις επόμενες εβδομάδες για να προωθήσουμε την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Εμένα με ενδιαφέρει η Κομισιόν να λάβει υπόψη και την κατεύθυνση την οποία υποδεικνύει το Κοινοβούλιο και ποια είναι η σκέψη του Κοινοβουλίου να μπορεί να το λάβει υπόψη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα με την έκθεση αυτή να δώσω μια πολιτική έκφραση των θέσεών μας η οποία θα επηρεάσει και τις κατευθύνσεις της Κομισιόν Μπορεί να είναι επαρκή οι ρυθμίσει που υπάρχουν τώρα, αλλά ίσω χρειάζεται η Κομισιόν να σκεφτεί για περαιτέρω ρυθμίσει για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση ή να διατηρήσει την ισότητα του ανταγωνισμού όταν έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση των κλασικών παρόχων και των νέων μορφών παρόχων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς για, που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση και δεσμεύομαι να κάνω και μια ευρύτερη παρουσίαση γιατί πρέπει να μπορέσει κανείς να δει πώς θα είναι στην πραγματικότητα αυτή η υβριδική τηλεόραση και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μια πιο εποπτική θα προσπαθήσω να το οργανώσω αυτό και θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορούν να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από εσά για να το δουν με, με τα βαΐων και κλάδων, με χρώματα και ήχους τι έχει να μας προσφέρει η νέα υβριδική τηλεόραση και να σκεφτούμε καλύτερα σε ποια σημεία θα πρέπει να παρέμβουμε και να εκπονήσουμε και νέες μορφές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ Πέτρα. Το Φεβρουάριο λοιπόν θα έχουμε το έγγραφο εργασία σου, αλλά σίγουρα θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψη για τα θέματα αυτά και ενδεχομένω να έχουμε κάποιες προτάσεις που θα μπορέσουμε να τις προωθήσουμε μαζί σου. Αυτά. Κλείνει λοιπόν η συνεδρία μας σήμερα και περνάμε στη συνεδρία των συντονιστών. Ναι. Short. Short.